να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος, λίγη εδώ συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση αύριο 12 Μαΐου 2011 από τις 9 ως τη 1 και από τις 3 ως τις 5 είναι διαθέσιμη η ημερήσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λίγη η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ.